9 και 2 η ώρα, νομίζω καλά είναι να αρχίσουμε. Πρώτο θέμα στην ημερησία διάταξη, έγκρισή της. Δεν ξέρω αν έχετε τίποτα αιτήματα για τροποποίηση της ημερησίας διάταξης. Όχι. Εγκρίνεται. Δεύτερο, έγκριση των πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων με τη γνωστή διαδικασία. Εάν δεν ε, υποβάλει κανείς αίτημα τροποποίησης ή απόρριψης κάποιου σημείου των πρακτικών θα θεωρηθούν εγκεκριμένα ε, μέχρι το τέλος της συνεδρίας. Για τη σημερινή συγκεκριμένη συνεδρίαση βεβαίως έχουμε ε, ηλεκτρονικά πρακτικά και έχουμε βάλει και μια ημερομηνία για την έγκριση για ότι στο προσεχές μέλλον δεν θα έχουμε κοινή συνεδρίαση άλλη των δύο επιτροπών μας, ΙΝΤΑ και ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ. Σημείο τρίτο. Ανακοινώσεις του Προέδρου. έχουμε δύο Προέδρους. Καλωσορίζω και τη συνάδελφο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών. Και συμφωνήσαμε να σας κάνουμε δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη ανακοινώτηση. Ω συνήθω η σημερινή συνεδρίαση μεταδίδεται απευθεία στο διαδίκτυο. Καλώς ορίσατε. Ε, οι οπαδοί του υπολογιστή και της τηλεόραση ανά την Ευρώπη. Επίση υπάρχει και ένα e-meeting ε, που μπορείτε να έχετε πρόσβαση όλοι οι βουλευτές ε, ε, στα έγγραφα και οι ενδιαφερόμενοι βοηθοί και έρχομαι αμέσω στο σημείο 4 και δίνω το λόγο στην Συμπροεδρόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε όλοι. Βρισκόμαστε εδώ τώρα για να ψηφίσουμε την έκθεση ε, που αφορά την εισαγωγή των πολιτιστικών αγαθών. Πριν ξεκινήσουμε ωστόσο την ψηφοφορία θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους εισηγητές. Στην κυρία Μόσχα και ο κύριο Ντάλτον θέλουν να κάνουν κάποια δήλωση. Ευχαριστώ. Πριν από την ψηφοφορία ήθελα να παρουσιάσω τη θέση μου. Θα δείτε ότι στη λίστα ψηφοφοριών δεν υπάρχουν συστασει του συνεισηγητή. Αυτό διότι σε μεγάλο βαθμό καταφέραμε να βρούμε συμφωνία για μεγάλο κομμάτι του κειμένου. Και έχουμε δημιουργήσει μια κοινή θέση που καλύπτει τα βασικά ζητήματα. Δυστυχώ, όσον αφορά τα τελευταία βήματα, δεν είχαμε τι ίδιε εμπειρίε. Και θεωρώ ότι το κείμενο αυτό δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Σημαντικά στοιχεία που είναι κλειδί για την υλοποίηση τη πρόταση δυστυχώ δεν είναι απολύτω έτοιμα. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτη και προβληματισμό. Αντιθέτω, ε, προς δική μου δυσαρέσκεια οι τελικοί συμβιβασμοί μας εστάλησαν από τους συζητητές με email μετά από μια τελευταία συνάντηση όπου κάποιες προτάσεις μπήκαν στο ράφι. Εγώ δεν συμφώνησα με κάποιες προτάσεις. Ε, θεωρώ ότι χρειάζονται περισσότερη μελέτη. Τώρα λυπάμαι. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε μια ε, συνεδρία συσκιωδών την πράσινη εβδομάδα ή την ομάδα της Ολομέλειας πριν λόγω προβλημάτων από πλευρά μου και από πλευρά κυρία Μόσκα. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο ότι έκτοτε όμως ε, θεώρησαν ότι ήμουν ε, κάποιος ε, συνεισηγητή που δεν μπορούσαν να μην λάβουν υπόψη. Ο σκιώδης Εγώ εκπροσωπώ την Επιτροπή ΙΜΚΟ και θεωρώ ότι η μεταχείριση αυτή δεν ήταν σωστή στην παρούσα φάση. Και ήθελα αυτό να γραφτεί στα πρακτικά, κυρία Πρόεδρε. Οπότε δεν προτείνω να εγκρίνουμε αυτές ε, τις ε, συμβιβαστικές Ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή όχι, δεν έχουν τηρηθεί οι κανόνε και οι πρακτικέ. Αποτελεί έλλειψη σεβασμού προ το άτομό μου και προ ε, την επιτροπή που εκπροσωπώ τώρα. Ξέρω ότι πάμε προ το τέλο τη θητεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μισοτελειωμένα πράγματα ή να υποβάλουμε προτάσει με τι οποίε διαφωνεί και ποιο από του συνεισηγητέ. Εγώ ως υπεύθυνο άνθρωπος δεν θα σταθώ ε, εμπόδιο στην έγκριση της απόφασης, αλλά θέλω να πω ότι ο συνεισηγητής και κεντρικό, με τον κεντρικό μου ρόλο στην κοινοβουλευτική διαδικασία θεωρώ ότι έχω απογοητευτεί. Γίνεται εσπευσμένα αυτή η διαδικασία και εγώ δεν συμφωνώ καθόλου και συνιστώ να το καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κρίμα που έγιναν ε, έτσι οι διαδικασίες. Δεν ξέρω αν η συγκεκριτή θέλει να κάνει... Να... Και θέλει να, κάνει κάτι, να πει κάτι. Ας προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Λοιπόν, έχουμε συμβιβαστική εκτός μικροφώνου, μιλήτρα. Όπως φαίνεται θα πρέπει να κάνουμε μια δοκιμή πρώτα απ' όλα. Να σας θυμίσω ότι είναι πόσο όμορφη η μέρα είναι σήμερα. Θα ψηφίσουμε για το κατά πόσο είναι μια όμορφη μέρα η σημερινή.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 They working. Yeah. Okay. Is it working, Roja? Yeah? Okay, perfect. Okay. Δουλεύει μια χαρά. So everybody is ready. So we start. Είμαστε όλοι έτοιμοι λοιπόν. Ξεκινά η ψηφοφορία. Συμβιβαστική τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Επιτροπή Πολιτισμού. Καλτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. συμβαστική τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 23. more Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Τροπολογία 188. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 189. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 189. πέρα ψηφοφορία απορρίπτεται. Συμβιβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29 υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 226. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Όχι. Καταπίπτει 27. Συμβιβαστική τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 228 δεν ψηφίζουμε και περνάμε στην συμβαστική 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 38. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 40 υπέρ. Α, ναι, 31 καταπίπτει. Συμβαστική 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 283 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται ελέγχουμε όμως ηλεκτρονικά την 283 We close the vote. And it is adopted. Εγκρίνεται. 284. Και αυτή καταπίπτει. Λάθος μου λέει ο πρόεδρος. 286 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 287 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τη 288. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 291. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 300. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 301. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 302. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. αποχές Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 47. Υπέρ. Κατά αποχές Συμβιβαστική 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 336 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβιβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 46. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Δεν βλέπω χέρια. Ξανά. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 27. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 357 υπέρ. Α, και αυτή καταπίπτει. Βέβαια, βέβαια, έχετε δίκιο. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Τροπολογία 50. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 360 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 360 παρακαλώ Κλείνουμε την ψηφοφορία εγκρίνεται πάμε στην 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 372 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 378 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 380 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 389 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 390 και 54 ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 392 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 393 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 394 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 395, 396 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνον, απορρίπτονται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 398 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 61 υπέρ, κατά, αποχές ε, ε, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές δύσκολο να ελέγξουμε την 62 ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Κλείνει η ψηφοφορία, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 402 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην 403 και 404 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε την τροπολογία 2. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 3 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 40 παρακαλώ.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 Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 14. Βλέπω στον καταλογό μου εδώ. Σωστά. Όχι.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 Πάμε στην... στα παραρτήματα. Συμβιβαστική 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και μετά πάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας και η έκθεση εγκρίνεται με την πλειοψηφία των 56 υπέρ, 4 κατά και 3 αποχές. And I would like to... Θα ήθελα... Θέλει κάποιος από τους εισηγητές να πει κάτι? Όχι. Α, ο κύριος Ντάλτον θέλει να πει κάτι. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα προηγουμένω, αλλά να πω ότι τώρα έχουμε μια θέση και όπως είπα και προηγουμένως ως ε, υπεύθυνο άνθρωπος ε, και ευρωβουλευτής δεν θα ε, φέρω κάποια αντίρρηση. Θα πάμε στη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και θα δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο πάλι στον συμπρόεδρό μου. Το μόνο που θέλω να κάνω εγώ είναι να ευχαριστήσω τους εισηγητές, τα μέλη και του διοργανωτέ τη κοινή αυτή συνεδρίασης, τη οποία κηρύσω και τη λήξη.